Να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλου. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρία τη Επιτροπή μα. Γκρίνουμε καταρχήν την ημερησία διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει. η ημερησία διάταξη γκρίνεται. Έγκριση των πρακτικών, συνεδρία στις 27 Μαρτίου, το δεύτερο σημείο και εδώ δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Σημείο 3. ανακοινώσει του Πρόεδρου, αγαπητοί συνάδελφοι, να υπενθυμίσω σε όλους ε, ότι έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε στη συζήτηση για τις προπτικές για τα δικαιώματα φύτευσης των αμπελώνων, για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που οργανώνεται από τη συνάδελφο Ελίζα Διάγκλε. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σήμερα στις 6.30 εδώ στην αίθουσα PHS 1α002 αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι web streamed. Αναμεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Κατόπιν, να καθοσλωσορίσω τον Επιτροπό Τζον Ντάλι, μέλο τη Επιτροπή Αρμόδια για την Υγεία και την Πολιτική Καταναλωτών. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε και πάλι εδώ. Κύριε Επίτροπο. υπάρχουν πολλέ πρωτοβουλίε που αφορούν την ε, υγεία και την ευημερία των ζώων. Έτσι λοιπόν, θα δώσω αμέσω ε, το λόγο στον κύριο Επίτροπο. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσει από του συντονιστέ και κατόπιν στα υπόλοιπα μέλη που θέλουν το λόγο. Έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής ε, γεωργίας για να, ως ε, Επίτροπος ε, Θεμάτων Υγείας και Καταναλωτών. τα θέματα τα οποία χειρίζομαι άπτονται των ενδιαφερόντων αυτής της Επιτροπής και είναι πολύ επίκυρα, ειδικά επειδή ορισμένα θέματα πρέπει να ολοκληρωθούν στο μέλλον. Δεν μπορώ βεβαίω να καλύψω τα πάντα, όλα τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Επίτροπή σα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, γι' αυτό θα επικεντρωθώ στο ουσιώδη. Και εν συνεχή θα είμαι στη διάθεσή σα για ερωτοαπαντήσει. Καταρχά, η ευζοία των ζώων και η υγεία των ζώων όσον αφορά την στρατηγική τη Ένωση για την προστασία και ευζοία των ζώων 2012-2015 καλωσορίζω την ε, συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιμένω ε, με μεγάλη ε, ικανοποίηση την, τα συμπεράσματα του σχεδίου έκθεσης της κυρίας Πόλσεν. Σας διαβεβαιώ αγαπητά μέλη ότι γνωρίζω ότι χρειάζεται μία ολοκληρωμένη εφαρμογή υλοποίηση των σημερινών νόμων και σημερινής νομοθεσίας για την ευζοία των ζώων και συμμερίζουμε τις απόψεις σας. Πρέπει η υλοποίηση, η εφαρμογή δηλαδή να γίνει περισσότερο σεβαστή και να είναι εξασφαλισμένη με συγκεκριμένα βήματα. Βεβαίω, η Επιτροπή γνωρίζει επίση ότι ενδέχεται να προκύψουν ε, επιπλέον δαπάνε ε, στου παραγωγού εφόσον εφαρμοστούν μέτρα βελτιωτικά τη ευζοία των ζώων. Γι' αυτό καταλαβαίνω απόλυτα ε, όσους θέλουν να δουν την Κομισιό να προτείνει νέες πρωτοβουλίες για τη μεταφορά, ε, τι γαλακτοφόρες αγελάδες ε, και τα κατοικίδια ζώα. Εγώ βεβαίως προτιμώ μια ολιστική προσέγγιση η οποία να εφαρμόζεται σε όλο το ζωικό βασίλειο με γενικούς μηχανισμούς. Πάντως, συμφωνώ γενικά ότι χρειάζεται μια νομοθεσία, ένα γενικό πλαίσιο νομοθεσίας για την ευζοία των ζώων, το οποίο να βασίζεται σε ένα δίκτυο κέντρων αναφοράς, το οποίο θα οικοδομηθεί βάσει των πιλωτικών προγραμμάτων, ε, τα οποία έχουν προάγει, έχει προάγει, έχει υποστηρίξει το Κοινοβούλιο, και ε, τα οποία, για τα οποία η Κομισιόν θα προκηρύξει μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Επίσης διαβεβαίω ότι θα λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Όσον αφορά τώρα την ευζοία των ζώων θα πρέπει να περιορίσουμε ε, το χρόνο μεταφοράς ε, σε 8 ώρες για τα ζώα που προορίζονται προς σφαγή. Έχω εξετάσει λοιπόν επί ενδελεχώς όλα τα στοιχεία της μεταφοράς των ζώων. Τα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάντε μεταφέρονται πάντοτε από τις μονάδες τους προς ε, τα σφαγεία και εκεί θα πρέπει να ακολουθούν τους πιο αυστηρούς ε, κανονισμούς. Θα πρέπει να ανταποκριθούν θα πρέπει να ε, ανταποκριθούμε λοιπόν στις οικονομίες κλίμακος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να μεταφέρονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις και βάσει των στοιχείων που έχουμε 60-70% ε, των ζώων μεταφέρονται σε σφαγεία τα οποία ε, και έτσι αναγκάζονται να είναι στο, στο καθοδόν πάνω από 8 ώρες. Καταλήγω λοιπόν ότι δεν είναι η στιγμή τώρα να προτείνουμε ε, αλλαγές στον κανονισμό μεταφορά ζώων και δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε αυτό. Ε, θα επικεντρώσουμε, πρέπει τα κράτη-μέλη να επικεντρώσουν την προσοχή τους, όπως επίσης και ο τομέας και η Κομισιόν, στην ε, σωστή εφαρμογή των τραχουσών διατάξεων και κανονισμών. Α, διαφορετικά θα διακινδυνεύσουμε μια διάσπαση και διάλυση του Διακοπή. Α, το μικρόφωνο χάθηκε. Παρακαλώ μικρόφωνο. Διαφορετικά θα κινδυνεύσουμε να διαλυθεί και να διασπαστεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην υλοποίηση, στην εφαρμογή και στην εφαρμογή, στην εισαγωγή ε, νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση του όλου πλαισίου μεταφράστων ζώων. Τώρα, υλοποίηση της οδηγίας ε, για την προστασία των και ε, ε, κινδυνεύει αυτή η οδηγία για την protection των χείρων να υποστεί την ίδια ε, μεταχείριση όπως η προηγούμενη οδηγία για την ευζοία των οτόκων ορνήθων. Η απαγόρευση ε, των μεμονωμένων μονάδων εγκατάσταση υιοθετήθηκε το 2001 με μια μεταβατική περίοδο 12 ετών για να δώσει τη δυνατότητα μιας ε, ε, ομαλής μεταφοράς αλλαγής του συστήματος από τις παραγωγικές μονάδες. Μόνο 16 μέλη, κράτη-μέλη ε, έχουν σεβαστεί και έχουν συμμορφωθεί με την ε, προθεσμία αυτή η 1 Πρώτη 2013. Μόνο 16. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ξεκάθαρη πλήρη εφαρμογή της οδηγίας μέχρι τη συμφωνηθεί σε προθεσμία. Το έχω πει αυτό στο Συμβούλιο και πιο πρόσφατα μάλιστα το δήλωσα στις 26 Απριλίου ενώπιον του Συμβουλίου. Η Κομισιόν δεν θα διστάσει να ξεκινήσει τις διαδικασίες προσφυγής σε περιπτώσει μη συμμόρφωση. Τώρα, η ε, ε, επισήμανση των ε, βοηδών. Σύμφωνα με τον τομέα θα πρέπει να όχι μόνο να επιβάλλουμε ένα σύστημα εφαρμόσιμο και εφικτό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, αλλά και να φροντίσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των παραγωγών και άλλων ενδιαφερμένων του τομέα of Η παρούσα, η τρέχουσα νομοθεσία στη ζωοτεχνική, η οποία ε, προωθεί το ελεύθερο εμπόριο, ε, έχει αποδειχθεί ωφέλιμη και λειτουργεί ικανοποιητικά, όμως πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την συνθήκη της Λισαβόνας και θα πρέπει 11 κάθετα νομικά κείμενα να, ε, συντονιστούν και να ευθυγραμμιστούν σε, μια πλουστευμένο, σε ένα πλουστευμένο κανονισμό. Η πρόταση, την οποία προβλέπω να υιοθεθεί το καλοκαίρι, έχει ως στόχο ακριβώς αυτή τη συνένωση και θα ενθαρρύνει την τροφή και παραγωγή ζώνη υψηλής γενετικής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει τη γενετική βιοπικιλότητα μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου όσον αφορά τα μέτρα προς υιοθέτηση θα υιοθετήσουμε ένα πακέτο τεσσάρων προτάσεων που θα αναφέρονται στην, ε, στην υγεία των ζώων και φυτών, στην, αναπαραγωγικό, αναπαραγωγικό φυτικό υλικό, ε, στις, στους ελέγχους και στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας. Να σας εξηγήσω ε, λίγο περισσότερο αυτές τις τέσσερις προτάσεις. Ε, ε, η νόμος, νομοθετική πράξη υγεία ζώων. Η πρόταση για ένα, μια νέα, ένα νέο τέτοιο νομοθετικό μέσο θα προβλέπει και την πρόληψη ασθενειών στα ζώα και επιδημιών. Θα ενσωματώνει, ορθολογίζει και απλουστεύει ε, ένα μεγάλο πακέτο νομοθεσίας και κανονισμών έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, ο φυτογειονομικός νόμος, φυτογειονομική νομοθεσία. Ο στόχος μιας νέας πρότασης είναι να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έναντι νέων ε, ζυζανίων, παρασίτων και να εξυγχρονίσουμε και ευθυγραμμίσουμε το τρέχον καθεστώς. Η παγκοσμιοποίηση και η κλιματική αλλαγή έχουν αυξήσει τους κινδύνους ε, και, και για τα φυτά και για τη φύση γενικά. Θα πρέπει να επισημαίνουμε έγκαιρα και να μπορούμε να εξα, εξαλείφουμε ε, τα νέα παράσιτα και έτσι να, ε, να εξοικονομούμε και δαπάνες αλλά και να αποφεύγουμε επίσης την πρόσθετη χρήση παρασιτοκτόνων. Ο νέος νόμος επίσης συμπληρώνει τη, τη στρατηγική της Η αναθεώρηση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού ε, ο στόχος είναι να εναρμονίσουμε και να απλοποιήσουμε 12 οδηγίες σε ένα νομοθετικό μέσο, σε ένα νόμο και να μειώσουμε το κόστος ε, το διοικητικό της εφαρμογής. Ε, Τέλος, μέσα στο πακέτο ε, οι έλεγχοι της αλληλείας θα αναθεωρηθούν για να μπορέσουμε να ορθολογήσουμε την τρέχουσα προσέγγιση. Όσον αφορά τον έλεγχο υπολοιμάτων και εισαγωγών, θα εισάγουμε και όλες τις απαραίτητες αλλαγές για να βελτιώσουμε ε, την αναθεώρηση των σπόρων, της υγείας των φυτών και των ζώων. Γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το πακέτο υγειονομικών μέτρων, το οποίο ενισχύει από το 2006 και έτσι θα παρουσιάσουμε προτάσεις μετά το καλοκαίρι με την αντίστοιχη μελέτη επιπτώσεων. Οι, πρότασεις, οι προτάσεις αυτές θα έχουν ως στόχο μικρές προσαρμογές σε διάφορους τομείς, απλούστευση, διευκρίνηση μείωση διοικητικού κόστους χωρίς να διακυβεύουν τα θεμελιώδη, τις θεμελιώδεις στόχους του πακέτου. Επίσης ε, θα ευθυγραμμίζουν την υγειονομική νομοθεσία με τις συνθήκες του Λισαβόνας. Ένα άλλο σημαντικό πρωτοβουλίο της Κομισιόν είναι η, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ε, και θα ε, δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εκφράσουν την άποψή τους και την προσέγγιση τους. Αν θέλουν να επιτρέψουν την, ε, εσοδία, την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων ή όχι. Η πρόταση αυτή έχει πλέον μπει σε μια καθοριστική φάση και ελπίζω να υπάρξει πολιτική συμφωνία μέσα στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος τον Ιούνιο. Ελπίζω θα συνεχίσουμε το πνεύμα της καλής συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου Κομισιών turning to another dossier which has proved more than a little difficult over the years honourable members will no doubt και έτσι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στη δεύτερη ανάγνωση νέα τρόφιμα ε, cloning Νέε τροφές Όπω ξέρετε, η Κομισιόν τώρα χειρίζεται το θέμα του cloning. Ξεχωριστά και θα υποβάλουμε μια νέα πρόταση το 2013 για την κλωνοποίηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να χειριστούμε χωριστά το θέμα της κλωνοποίησης από τα νέα τρόφιμα. Τα δύο αυτά ντοσία ξεχωριστά στις αρχές του 2013. Σας παρουσίασε λοιπόν με μια σύντομη ανασκόπηση των ντοσία των φακέλων που έχουμε στο τραπέζι μας και τα οποία μας αποσχολούν και <clears throat> τα οποία είναι λίγα επίκαιρα. Πιστεύω έντονα ότι θα παίξετε ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας των ε, θεσμικών οργάνων. Και γι' αυτό θα συνεργαστώ στενά μαζί σας για να εξασφαλίσουμε ότι οι ενέργειές μας θα είναι συντονισμένες και θα εξασφαλίσουμε η καλύτερη ζωή για τους ε, πολίτες μας. Και τώρα θα ήθελα με μεγάλη ευχαρίστηση να ακούσω τις απόψεις των μελών της Επιτροπής και να απαντήσω σε ερωτήσεις που τυχόν έχετε. Ευχαριστώ, αγαπητέ Επίτροπα να δώσουμε τώρα το λόγο στους συντονιστές ευθύς αμέσως. Έχουμε πάρα πολλούς που έχουν ζητήσει το λόγο. Ας ξεκινήσουμε τον Αλμπερντές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή μας και ευχαριστώ ιδιαίτερα εκ μέρους του ΕΛΚ για την πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε μαζί σας και ιδιαίτερα κάθε φορά που είχα ένα αίτημα, σα παρουσίασα ένα αίτημά μας, ε, αντιδράσατε, ενεργήσατε ταχύτατα και ανταποκριθήκατε ε, πολύ καλά και γρήγορα, το οποίο δεν συμβαίνει σε όλες τις γενικές διευθύνσεις. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στα συγκεκριμένα θέματα που αναφέρετε εσείς, αλλά θα ήθελα σήμερα να θίξω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα της περιφέρειάς μου. Όπως ξέρετε είμαι βαβαρός από την, από την περιοχή του Oberklaus και έχουμε 14.000 μικρές λίμνες. Είναι η πιο πλούσια ε, περιοχή, η πιο πολυπληθής περιοχή μικρών λιμνών όπου γίνεται και ψάρεμα και... Λόγω αυτής της ε, μικρής κλίμακας αλίας εμπίπτει στις διατάξεις της αλίας γενικά. Πρέπει όμως εμείς να βρούμε μία άλλη ρύθμιση λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων και θα σας καλούσα να επισκεφθείτε αυτή την περιοχή των λιμνών για να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί και ε, πώς αυτή, μία ασθένεια η οποία έχει τώρα θίξει τα ψάρια στις λίμνες αυτές δεν έχει καμία επίπτωση στις άλλες ασθένειες των ψαριών που καλύπτονται από τα γενικά θέματα αλίας και γι' αυτό πρέπει να γίνει ξεχωριστή μεταχείριση αυτής της επιδημίας. Είπατε ότι ε, επί το θέμα των σφαγίων τώρα, επί το θέμα των σφαγίων, όλο και περισσότερα σφαγεία κλείνουν. Και γι' αυτό οι μεταφορές γίνονται όλο και πιο μακρινές. Πρέπει όμως εμείς να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των ε, σφαγίων. Να μην επιμηκύνονται συνέχεια οι χρόνοι μεταφοράς των ζώων. Έχουμε δει σε τόσες πολλές περιοχές να κλείνει το ένα σφαγείο μετά το άλλο. Πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Κάποια λύση πρέπει να βρεθεί σε αυτό το πρόβλημα. Να μπορούν να επιβιώσουν αυτά τα σφαγεία έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βραχία μεταφορά των ζώων. Αυτά τα δύο ε, αιτήματα είχα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κατόπιν ο Λουίς και μετά ο Τζον Λάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε πίτροπε. Η έκθεση των ε, προτεραιοτήτων της Επιτροπής για τον επόμενο ε, χρόνο έχουν να αντιμετωπίσουν τι ανησυχίες μας. Περιμένουμε βέβαια να δούμε το περιεχόμενό τους, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της φυτογειονομικής νομοθεσίας. Γνωρίζουμε ότι οι απειλές για την Ευρώπη και είναι πάρα πολύ μεγάλε. μάλιστα και για του λόγου που αναφέρατε και μα ανησυχούν όλα αυτά και περιορίζουν την ε, ικανότητά μα. να ανταγωνιστούμε. Έτσι λοιπόν... Ε, Περιμένουμε από τον κύριο Επίτροπο να μας αναφέρει το περιεχόμενο των προτάσεων αυτών και θα ήθελα να σας πω πόση σημασία δίνουμε στην στο ζήτημα αυτό και στην αναγκαιότητα να προχωρήσουμε όσο δυνατόν ταχύτερα. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί, θα περάσω σε κάποιες μεγαλύτερες λεπτομέρειες, που έχουν να κάνουν ε, με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και τα υπολείμματά τους ε, ε, στα μεταποιημένα προϊόντα. Έχουμε διάφορους εισαγωγές που μας λένε ότι είναι αδύνατον να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα υπολείμματα σε προϊόντα για την διατροφή των ανθρώπων ή για την τροφή των ζώων. Έτσι λοιπόν μας λένε ότι είναι αδύνατον να το ξεχωρίσουν ανεξάρτητα από τον προορισμό του. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξεκαθαρίσει η Κομισιόν και θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν αν σκοπεύει να κάνει κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω έχει να κάνει με τις ποικιλίε καπνού που παραγόνται στην Ευρώπη και που θεωρούνται ε, βλαβερές για την υγεία. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν αν σκοπεύει να αναθεωρήσει την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Και, κύριε Επίτροπε, έχω και ένα σύνολο άλλων ερωτήσεων, αλλά αυτή τη στιγμή αυτές θα θέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λουίς Τζορτζ Λάιον και κατόπιν Τζιμ Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Επίτροπο και να το συγχαρώ για το ότι έχει πολύ καλές ε, σχέσεις συνεργασίας με αυτή την Επιτροπή. Το εκτιμούμε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό για μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά θεμάτων που θίξατε και να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχήν, για την στρατηγική για την ευημερία των ζώων. Υποστηρίζω πλήρως την άποψή σας ότι η επιβολή είναι το θέμα κλειδί, το βασικό ζήτημα ότι δεν θέλουμε μεγαλύτερη νομοθεσία, θέλουμε να εφαρμόζεται ορθά η νομοθεσία έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η νομοθεσία για την ευζοία των ζώων ε, τη θέση εφαρμογή ορθά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση τώρα με τα όσα αναφέρατε, μπορώ να υποστηρίξω την άποψή σας ότι ε, η επιβολή της νομοθεσίας είναι πολύ πιο σημαντική. Σε ένα σενάριο στη Σκωτία θα σήμαινε ότι πάρα πολλοί ε, κτηνοτρόφοι στις νήσους δεν θα μπορούσαν να μεταφέρουν το ζώο τους στις αγορές. Θα πρέπει πάντοτε να σεβόμαστε την επιστήμη σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν όμως κάποια επιστημονικά στοιχεία, αλλά πρέπει πάντοτε να δούμε τι λένε οι επιστήμονες και να λαμβάνουμε αποφάσεις. Ε, ε, είπατε τώρα ότι 16 κράτη-μέλη θα σέβονται ε, την οδηγία για τους χειρούς μέχρι τα τέλη του έτους. Όμως ε, τα κράτη-μέλη που δεν θα σεβαστούν την οδηγία θα προσφύγετε κατά αυτό στο δικαστήριο. Ε, θέλουμε... Είδαμε ότι και οι λιανέμποροι ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για το θέμα αυτό και η δική σας ε, υπηρεσία έκανε, υλοποίησε μια απειλή για προσφυγή στη δικαιοσύνη. θα επιταχύνεται με αυτόν τον τρόπο αυτή τη διαδικασία και ίσως κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία έτσι ώστε οι λιανέμποροι να μην ε, αποθηκεύουν ε, μόνο ε, κρέας ε, που έχει υπάρξει βάση προτύπων. Τώρα, για τις οτόκες όρνηθες αναφέρατε ε, κάποια δράση που αναλαμβάνετε. Μπορείτε να μας πείτε τι αποτελέσματα αναμένουμε στα κράτη-μέλη, πότε θα σέβονται πληρώς την νομοθεσία, μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για τα δύο τελευταία θέματα που αναφέρατε, ε, για την ε, πολιτική συμφωνία, για το θέμα της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων, ε, για το να επιτευχθεί μια συμφωνία τον Ιούνιο. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ομοθεσία αυτή, πότε θα εφαρμοστεί και σε σχέση με την πρόταση για τα νέα τρόφιμα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το να παρουσιάσετε μια νομοθετική πρόταση γι' αυτό. Ξέρω ότι είστε σε διαδικασία διαβούλευσης αυτή τη στιγμή, αλλά θα υπάρχει μια νομοθεσία που θα έρθει στο Κοινοβούλιο πριν τη λήξη αυτής της θητείας το 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζιμ Νίκολσον. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Επίτροπο με τη σειρά μου. Είπατε ξεκάθαρα ότι ακολουθούν αλλαγές, ε, είναι πολλοί οι τομείς όπου θα υπάρξουν αλλαγές. Θα συμφωνήσω με τον Τζο Λάινε δεν μπορούμε να έχουμε έναν ουρανοκατέβατο αριθμό που θα εφαρμόζουμε σε όλες τις περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους καλύτερους μηχανισμούς και τα καλύτερα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας για να επιτύχουμε την ε, ε, ευημερία των ζώων που επιθυμούμε και φυσικά να δικαιολογείται η δράση μας από τα επιστημονικά στοιχεία. Δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω αυτή τη θέση. Είπατε και το ξέρουμε όλοι ότι ε, έχουμε 16 κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται με τα χειροστάσια, τα μεμονωμένα ατομικά χειροστάσια. Ε, πέρσι, όταν ασχολούμαστε με τις όρνηθες και τους κλωβούς, ε, είχαμε το ίδιο θέμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ε, εξετάζουμε τα θέματα από οπτικής γωνίας ευζήν των ζώων ε, εκτρέφουμε αυτά τα ζώα και παράγουμε ε, χάρη σε αυτά τα τρόφιμα και θέλουμε υψηλότερα πρότυπα. Μα ποιος ε, προσπαθεί να παρεμποδίσει τις προσπάθειές μας και να αλλάξει την κατάσταση ε, ενώ έχουν ήδη ε, αποφασίσει κάποια κράτη-μέλη, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε επαφή με, αυτή, με την πραγματικότητα. Ε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε απαγορεύσεις διαρκώς που δεν εφαρμόζονται. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία. Σωστή εφαρμογή Νομοθεσία ε, χρειαζόμαστε και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ε, και τώρα και στο μέλλον. Ε, Κυρίω σε αυτή την περίοδο όπου οι κυβερνήσει των κρατών μελών δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν τα απαιτούμενα κονδύλια. Το ίδιο και οι γεωργοί, το ίδιο και οι εκτροφεί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να συμμορφωθούν με τα πρότυπα. Και τότε η δουλειά μα είναι να μεριμνήσουμε ώστε αυτά που κάνουμε να είναι και εφαρμόσιμα. Κάτι άλλο που είπε ο Λουίς Κάπουλα Σάντος ε, σε σχέση με τα, τους γενετικά, ε, τα τρόφιμα με γενετικά τροπημένους οργανισμούς που εισάγονται στο Ρότερνταμ. Ε, όσοι εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φοβούνται διότι μπορεί να απορρίψει κάποιος τα εμπορεύματά τους στα λιμάνια. Ξέρετε, δεν πρόκειται να συμβαίνει αυτό στο μέλλον. Ναι. Δεν ναι, μπορούμε εμεί να σταματήσουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Είναι σαν να αυτό πυροβολούμαστε όταν εγκρίνουμε νομοθεσίε που δεν μπορούμε καν να εφαρμόσουμε. Ευχαριστούμε, Τζιμ, Μάρτιν Όσλι και μετά Άγνιο. Ναι, κύριε Επίτροπο, από τη δική μας πλευρά χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ. Και θα συνεχίσω μετά από αυτά που είπε ο Νίκ. Η, τα νέα κατόφια ανοχής στις εισαγωγές τροφίμων. Ε, στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, μια τέτοια πρόταση είναι πολύ επικίνδυνη διότι πολλές χώρες δεν επιτρέπουν την εισαγωγή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν έντονες ε, συζητήσεις ε, και θα ήθελα να ξέρω μεγαλύτερες, ε, περισσότερες λεπτομέρειες τι προτείνετε, πότε ακριβώς προτείνετε και επίσης στους ε, σπόρους ε, φύτευσης ε, θα ήθελε και εκεί να ξέρω τα μέτρα, καινούργια μέτρα ανοχής διότι και εκεί θα πρέπει να εφαρμόσουμε μηδενική ανοχή, μηδενικό ποσοστό ανοχής στους σπόρους φύτευσης. Διαφορετικά θα έχουμε μεγάλες αντιδράσεις από τους παραγωγούς. Όσον αφορά τώρα την νομοθεσία γενετικής, η πρόταση της Κομισιόν δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία εμείς ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία. Οπότε πώς να ερμηνεύσουμε το μήνυμά σας, ότι δεν λαμβάνετε υπόψη ε, τις προτάσεις μας ε, για την ε, γενετική νομοθεσία. Δεν λέω ότι πολλά θέματα επιδανικής προεδρίας δεν ρυθμίστηκαν, αλλά παρόλα αυτά δεν συμπίπτουν οι απόψεις μας. Όσον αφορά τώρα τη νέα πρόταση που λέτε για τα νέα τρόφιμα και κλωνοποίηση, ε, μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα κατά πόσο θα προσεγγίσετε τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Ε, ξέρετε ότι απέτυχαν διαβουλεύσεις που κάναμε διότι η Κομισιόν δεν ήθελε να επιτρέψει μία ρύθμιση εισαγωγών για τις επερχόμενες ε, γενναίες. Τι εννοείται τώρα, θα αναθεωρήσετε τις παλαιότερες ε, προτάσεις ή θα προβάλλετε εντελώς καινούριε. Όσον αφορά τώρα τη χρήση αντιβιωτικών, δεν ξέρω αν είσαστε ενήμερος για τις ε, έρευνες, για τις εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν στη Γερμανία υπάρχουν, ε, υπάρχει μεγάλη ε, χρήση αντιβιωτικών. Τώρα, ορισμένες φορές χρειάζεται χρήση για δύο μέρες μόνο. Άλλες φορές στα, <clears throat> στα ζώα που θυλάζουν χρειάζεται περισσότερο. Αναρωτιέμαι λοιπόν να είσαστε ενήμερος για το αν γίνεται κατάχρηση, υπερβολική χρήση δηλαδή αντιβιωτικών. Πριν από έξι μήνες έχω αποστείλει μία επιστολή στην υπηρεσία, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Τώρα για την φυτοϊγειονομική προστασία έχετε υπόψη σα τα είδη τα οποία θα πρέπει να προστατευτούν, παραδείγματος χάρη σε περιπτώσεις ξηρασίας. Εκεί όμως ε, το μεγάλο κίνδυνο που διαβλέπω είναι ότι χάνουμε συνέχεια ήδη και έτσι θίγεται βεβαίως η βιοπικιλία, η βιοπικιλότητα. Ποια μέτρα θα εφαρμόσετε για να εξασφαλίσουμε την, ε, και να εγγυηθούμε τη βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγνού. και κατόπιν θα κλείσουμε με τους ε, συντονιστές. Θα απαντήσει ο κύριος Επίτροπος και θα συνεχίσουμε. Αν ε, δεν ξεκινήσω τη μικρή μου συνεισφορά με το να σας συγχαρώ, πιστεύω θα με κατανοήσετε, γιατί δυσκολεύομαι να το κάνω σε οποιοδήποτε επιτρόπο, αλλά δεν έχω κάτι προσωπικό απέναντί σας. Θα ήθελα Ήθελα να μιλήσω για τα ατομικά χειροστάσια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 16 κράτη λένε ότι θα σέβονται ε, την ομοθεσία μέχρι ε, τη δεύτερη παρουσία. Όμως ε, το θέμα είναι πώς θα συμμορφωθούν επειδή έχουν τη συγκεκριμένη τομέα. Γιατί εδώ βλέπουμε μεγάλο μέρες σε επίπεδα παραγωγής. Πρέπει να ρωτήσουμε αν κάποιες χώρες λένε απλά στην Κομισιόν αυτά που θέλει να ακούσει και προσπαθούν να εξαγοράσουν χρόνο. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπε χώρε. Είναι ντροπιαστικό ότι ούτε καν προσποιούνται ότι συμμορφούνται ή δεν συζητούν καθόλου το θέμα σε ορισμένε περιπτώσει. Πώ ε, ε, μπορούν να ανταγωνιστούν οι Βρετανοί που ε, συμμορφώνονται στην ενιαία αγορά. Η Κομισιόν ορισμενε περιπτωσει πω μπορουν να διαχειριστεί την κατάσταση γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούμε στο να εισάγουμε μεγάλες ποσότητες κρουκρες από ε, άλλες χώρες και καθώς μιλώ Ισπανία εισάγει τώρα αυγά από το Μεξικό καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει απαγόρευση αυτών των κλοβών για τις ε, οτόκες ε, όρνηθες. Για την μεταφορά των ζώων υπάρχει επαρκής νομοθεσία ε, εδώ, απλώς πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Και θα ήθελα, ενώ έχω την ικανότητα να ακούσουμε την Μανιχασμίνη να μας πει, μπορώ να σας πω ότι καμία ποικιλία δεν εξαφανίζονται, πάντοτε διατηρούν το πόθεμα ή κτηνοτρόφοι, γιατί μπορεί να χρειαστούν ε, ξανά ε, κάποια συγκεκριμένη γενετική ιδιοκτησία. Ποτέ δεν ξέρουν πότε θα τη χρειαστούν και τη διατηρούν. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πετρίπο για να απαντήσει στους συντονιστέ ε, και κατόπιν θα συνεχίσουμε. Κύριε Πίτροπε. thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω όλα τα επιμέρους σημεία που έγιναν οι συντονιστές. Ε, πρώτον, ο κύριος Ντέσσαν. Ε, σχετικά με τους Κυπρίνους ε, στις λιμνούλες ε, που έχετε και τις νόσους που πλήττουν τους Κυπρίνους. Κοιτάξτε, αναθεωρείται τώρα η νομοθεσία στα πλαίσια της γενικότερης νομοθεσίας για το ευζήν των ζώων σε σχέση με τα σφαγεία, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Όσα περισσότερα ε, σφαγεία κλείσουν, τόσο περισσότερα ζώα θα κινδυνεύουν. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι στην Ευρώπη και δεχόμαστε επικρίσεις ε, κατά της ε, νομοθεσίας, ε, δηλαδή ισχυρίζονται πολλοί ότι λόγω της νομοθεσίας δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι ως προς τα υγειονομικά μέτρα ε, που δίνανται να αναλάβουν τα κράτη-μέλη προβλέπεται μεγάλη ευελιξία μέσα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην όμως δεν χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη την ευελιξία που είναι σαφώς ενσωματωμένη μέσα στα νομοθετήματα και μας λένε ότι εξαιτία σας ε, έχουμε όλες αυτές ε, τις αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βασική μέρημνά μας είναι να εξηγήσουμε ότι το Κοινοβούλιο και όχι μόνο και το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ιδίως συνομοθέτες, δηλαδή και η Επιτροπή προσπαθούν να καλύψουν ναι, τις ε, διαφορετικές ανάγκες μικρότερων και μεγαλύτερων σφαγίων. Ναι. Ε, πρόσφατα ε, ήμουνα με τον Τάρσιαν Τσόλος σε μια διάσκεψη για το slow food, την αργή τροφή και μας μίλανε τους γεωργούς στα βουνά της Αυστρίας που θα ήθελαν ουσιαστικά να εμπορευθούν ε, προϊόντα, τρόφιμα που προέρχονται από ζώα που εκτρέφουν οι ίδιοι και ξέρετε ότι η ευελιξία υπάρχει, γίνεται αυτό. Ε, φυσικά τα θέματα υγιεινής και δημόσιας υγείας έχουν καθοριστική σημασία και πρέπει να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να ε, ε, εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες αναπερίσταση. Ε, τώρα θα απαντήσω στον Λουίς Κάπουλα Σάντος. Δίκιο έχετε, δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες διότι εκπονούνται νομοθετικέ προτάσει και η αξιολόγηση αντικτύπου γίνεται ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Όμω θα υποσχεθώ ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για μία συγκεκριμένη ειδική πρόταση θα συναντηθώ μαζί του και θα συζητήσω ε, για να έχω και τη συμβολή σα προτού καταθέσουμε και οριστικοποιήσουμε την ε, πρότασή μας. Δεν θα συμφωνήσουμε απαραίτητα σε όλα, αλλά τουλάχιστον θα έχει προηγηθεί συζήτηση και θα είμαι ιδιαίτερα ιδιαίτερα δεκτικός, ε, ο συνήθως άλλωστε, ε, στα σχόλιά σας. Για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, πολλοί σχολίασαν αυτό το θέμα, κυρίως όταν ε, μιλάμε για την χαμηλή παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αλλάξαμε τον τρόπο μέτρησης και τους σχετικούς κανόνες πριν από λίγους μήνες ε, για τις ε, εισαγωγές ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το σύστημα ισχύει εδώ και αρκετούς μήνες και αυτή τη στιγμή αναλύουμε τις επιπτώσεις ή τα οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν ε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ε, φαίνεται ότι βαίνουν όλα αισίως ε, και υπενθυμίζω σε όλους ότι η τροποποίηση του μηχανισμού μέτρησης εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο και τώρα εξετάζουμε το ενδεχόμενο να επεκτείνουμε αυτήν την, ε, ε, αυτό το νέο μηχανισμό μέτρησης ε, και στα τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση. Γενικώ έχουμε μηδενική ανοχή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά υπάρχουν διαφορές ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης. Υπάρχει τρόπος να έχουμε ένα συνεκτικό, μια συνεκτική μέθοδο μέτρησης για τους σπόρους. Προς το παρόν δεν εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή προτείνουμε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε για τις ζωοτροφές για τα εισαγόμενα τρόφιμα. Τώρα, για τον καπνό, ναι, όντως ε, προβλέπουμε αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού Οι επικεφαλείς μου μου λένε ότι είναι ύψιστη σημασία στο ζήτημα γιατί ο καπνός είναι ο βασικός φωνιάς που έχουμε ε, στην σημερινή κοινωνία αλλά θα ήθελα να σας καθησυχάσω για το εξή τουλάχιστον. Ε, τα πρόσθετα και οι διάφορες πρόσθετες ουσίες ε, είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί ε, και θέλουμε να σχεδιάσουμε μια δράση ούτως ώστε να ταξινομούμε τα, τις αρωματικές ουσίες και γενικότερα τις πρόσθετες ουσίες. Όμως ε, θέλουμε τα προϊόντα του καπνού να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά και προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία, ούτως ώστε να μην υπάρξουν αρνητικέ επιπτώσεις για τα προϊόντα του καπνού. Η διαδικασία της αξιολόγησης αντικτύπου που τώρα ακολουθούμε είναι ιδιαίτερα επαχθής. Φυσικά θα περάσει και από το Κοινοβούλιο και θα έχετε κάθε δυνατότητα να συζητήσετε κι εσείς όλες τις προτάσεις που θα ε, καταθέσουμε. Από όσο γνωρίζω πάντως δεν θα επηρεαστεί ο τομέας αυτός ε, του, της καπνοπαραγωγής παρά μόνο βεβαίως ως προς την κατανάλωση που ελπίζουμε να μειωθεί ε, δεν μπορώ παρά να ομολογήσω αυτό το πραγματικό ουσιαστικό στόχο μας. Σε σχέση με τον κύριο Λάινε πάλι θα συμφωνήσω 100% και δεν είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Όντω 100% εφαρμογή. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε και επιστημονική βάση για όλα τα στοιχεία. Θα λάβω ένα εκατομμύριο υπογραφέ ε, παραδείγματο χάρη την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τον όρο, το ωράριο μεταφορά που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8ωρο. Εντάξει, καταλαβαίνω τι ανησυχίε που εκφράζεται. Καταλαβαίνω ότι γίνονται καταχρήσεις, όμως ε, θα έπρεπε ε, όλοι από κοινού να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση. Και όπως σας είπα στην ανακτήρια ομιλία μου, αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι ε, να βρω έναν τρόπο ούτως ώστε να εφαρμόσουμε όλες τις διατάξεις περί μεταφοράς ζώων με ορθό τρόπο. Έχουμε τους κανονισμούς, σήμερα έχουμε και την τεχνολογία, ε, λοιπόν ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την σημερινή τεχνολογία για να κατοχυρώσουμε ότι ε, οι κανονισμοί θα εφαρμόζονται. Και το παράδειγμα που σας δίνω είναι ότι στο iPad μου σήμερα το, ε, έχω τη δυνατότητα να βλέπω όλα τα αεροσκάφη που πετούν αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει και μας επιτρέπει να ιχνηλατούμε, να παρακολουθούμε οποιαδήποτε μετακίνηση Μπορούμε λοιπόν ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα και όποιος ε, κάνει μία παρατυπία μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα σήμανσης Να ξέρετε όμως ότι η λύση σίγουρα δεν μπορεί να περάσει μόνο μέσα από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη επίσης πρέπει να δεχθούν οποιαδήποτε λύση προκρίνουμε. Ε, και χρειαζόμαστε ένα μάλλον κεντρικό σύστημα διότι είναι διασυνοριακό ε, το θέμα και η μετακίνηση ε, σχετικά με, τις, με τους χείρους θα συμφωνήσουμε με τους γεωργούς τόσο ώστε να έχουμε την σωστή εφαρμογή θεωρούμε ότι οι εκτροφείς μπορούν να μας βοηθήσουν επί τόπου ε, ούτως ώστε να εφαρμοστεί σωστά αυτός ο κανονισμός για τις χειρομητέρες. Τι κάνει ε, η Επιτροπή από πλευράς της ε, χρησιμοποιούμε, αξιοποιούμε στο έπακρον την νομοθεσία που έχουμε και αυτή η στάση που τηρούμε ορισμένε φορέ να είμαστε υπερβολικά αυστηροί με τα κράτη-μέλη έχει το εξή αποτέλεσμα. Σα δίνω ένα παράδειγμα. Ε, δεν θέλουμε να παραταθεί μία προθεσμία. Και μένετε ε, στη θέση σας. Ξέρετε τι σημαίνει. Δεν έρχονται καν να ζητήσουν παράταση προθεσμιών οι ενδιαφερόμενοι γιατί ξέρουν ότι θα τους το αρνηθούμε. Και ξέρω τώρα ότι ασχολούνται πολύ περισσότερο με τη συμμόρφωση και αυτό επιθυμούμε. Ακόμη και για τα χρηματοδοτικά ζητήματα του ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία και τα διάφορα διαθέσιμα ταμεία και να ε, συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία αλλαγή ε, για να συμμορφωθούν οι οτόκε όρνηθε τώρα. Έχουμε ε, μηνιαίω σύσκεψη με του εθνικού εμπειρογνώμονε και η θέση μας ε, ως, ε, προς το παρόν έχει ως εξής. Μέχρι το πέρας του τρέχοντος ε, θα έχουμε επιτύχει πλήρη συμμόρφωση. Αυτό συνάγουμε από τις τοποθετήσεις των κρατών μελών. Δεν ξέρω αν μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε ή αν τα εννοούν. Δεν μπορώ να... Την τηλεπάθεια δεν την κατέχω ακόμη. Ε, Όμω πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα των κρατών μελών, διότι ακόμη και αν μα λένε ψέματα τώρα, σε τρία ή τέσσερι μήνε ε, θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και είναι τίθεται και ζήτημα αξιοπιστία. Ε, πραγματικά πιστεύω ότι κάνουν σοβαρέ προσπάθειε για να συμμορφωθούν και μα διαβιβάζουν ορθέ πληροφορίε και στοιχεία. Θα συμφωνήσω πολύ δε και με τον κύριο Νίκολσον για το θέμα των μεταφορών, ότι πρέπει να ε, ε, είναι στοιχειοθετημένα επιστημονικά τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για να αποφασίζουμε και όλοι ε, ε το δημοφιλές πόρο τώρα τη σήμερα ημέρα είναι όλοι, όλα να τα ρίχνουμε στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής. Μπορεί να μην ε, φτάνουμε στον τόσο ψηλό πύχη που έχουν θέσει όλοι οι υπόλοιποι, αλλά πάντως ε, κάνουν, βάζουμε τα δυνατά μας για να ε, επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση. και για να καλύψουμε τις ανησυχίες των πολιτών, των καταναλωτών, των εκπροσώπων των εκτροφέων και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα προβλήματα όλων και κυρίως ε, να βρούμε μία συμβαστική λύση με την οποία μπορούμε να εργαστούμε στο μέλλον και να την εφαρμόσουμε. Σε σχέση τώρα με ε, τους γενικά τροπημένους οργανισμούς και τη θέση του κυρίου Χάουσλινγκ, ε, είναι προφανές ότι θα ακολουθήσει συνδιαλλαγή και ελπίζω να βρούμε κοινό παρονομαστή με το Συμβούλιο ως προς μία δεχόμενη πρακτική ε, λύση, ε, μάλλον μια λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ε, στην πράξη. Θα πιέσουμε για να επιλεχθεί μια λογική λύση. Όταν είδαμε τη θέση του Κοινοβουλίου, εμείς απαντήσαμε πως συμφωνούμε με την πλειοψηφία των θέσεων του Κοινοβουλίου και ότι θα στηρίζαμε το Κοινοβούλιο στη συνδιαλλαγή. Τώρα το Συμβούλιο καταθέτει προτάσεις με κάποια νέα στοιχεία και πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε και με τις επιτροπές και με το σύνολο του Κοινοβουλίου. Ως προς την κλωνοποίηση θα έλεγα ε, ότι η θέση μου, όπως εξάλλου σας υποσχέθηκα, για τις συζητήσεις για τα νέα τρόφιμα ότι θα είναι εντελώ αυτόνομο το θέμα ε, της κλωνοποίησης και θα καταθέσω μια ανεξάρτητη ξεχωριστή ε, πρόταση ε, σε σχέση με τα νέα τρόφιμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα πάω να τους ρωτήσω ακριβώς πώς θέλουν να προχωρήσουμε. Εγώ τίποτα δεν θέλω να προδικάσω. Αυτό που επιθυμώ και αυτό που σας συστήνω είναι ευθύ αμέσω να συνεχίσουμε με όλα τα νέα τρόφιμα αφαιρώντας μόνο το την κλωνοποίηση ίσως ε, ε, εξαιρουμένων κάποιων ρητρών διασφάλισης ε, που εκτάκτως θα υιοθετήσουμε. Η αξιολόγηση αντικτύπου ήδη γίνεται τώρα για την οδηγία κλωνοποίησης και η πρότασή μας θα ακολουθήσει για να συζητηθεί. Συμφωνώ μαζί σας πάντως ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία που ε, δεν θα περατωθεί. Και σήμερα γνωρίζω ότι άμα ε, επιχειρήσω και πάλι τα νέα τρόφιμα μαζί με την, ε, χωρίς την κλωνοποίηση θα σημειωθεί επιτυχία. Δεν μπορώ παρά να περιμένω το πράσινο φω ε, του Κοινοβουλίου για να προχωρήσω, για να είμαι σίγουρο. Αλλιώ, αν δεν μου δώσετε το OK για να προχωρήσω και για τα δύο θέματα, θα πρέπει να καταθέσω δύο διαφορετικέ προτάσει. Ε, για τα αντιβιωτικά στην, για τη χρήση του ε, στην γεωργία. Συμφωνώ, είναι εντελώ καταχρηστική αυτή η συμπεριφορά να χρησιμοποιούνται τι ούτω τρόπο δηλαδή τα αντιβιωτικά. Εάν είχατε παρακολουθήσει αυτά που λέγαμε όταν, εξαγγείλ, όταν δημοσιεύσαμε την ανακοίνωσή μας ε, για την ε, ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Είχα πει δημοσίως, επανειλημμένα κιόλας, πως το πρόβλημα με την αντοχή στα αντιβιωτικά είναι η κατάχρηση για κτηνιατρικούς σκοπούς και για θεραπευτικούς σκοπούς για τους ανθρώπους και στους δύο τομείς. Άρα θα πρέπει να δούμε αυτό που είπατε το 90% είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή ε, χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά ε, για τις... Ε, για διάφορες ζωονόσους, ε, κατά 90% και ε, οπωσδήποτε ένας κτηνίατρος ε, οφείλει να είναι παρόν όταν χορηγείται τέτοια αγωγή στο ζώο. τη στιγμή που χορηγείται συμβαίνει αυτό, πιστεύετε στις περισσότερες περιπτώσεις. οπωσδήποτε είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Άγνιου, νομίζω ότι τον έχω καλύψει με τις απαντήσεις που έδωσε μέχρι στιγμής θα καλυφθείτε πιστεύω από τις υπόλοιπες απαντήσεις μου ή θα εμπνευστείτε. Ευχαριστούμε για αυτές τις πρώτες απαντήσεις. Ε, πολλά υπόθηκαν. 13 άτομα έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο και κάποιοι ακόμη ζητούν το λόγο. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην χρονοτριβήσετε διαφορετικά. Δεν θα μπορέσει ο Επίτροπος να απαντήσει στο τέλος. Δεν κατόπιν καρόνα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε είχα ασκήσει έντονη κριτική στον Επιτροπό στο παρελθόν όταν ε, εδώ σε αυτήν την Επιτροπή μίλησε για την απαγόρευση των κλοβών. Δεν ε, θα εκνευριστώ και πάλι τόσο πολύ, απλώς ε, όταν μιλάμε για τους κλοβούς, για την ευημερία των χείρων ή για τη μεταφορά. Το, αυτό που μας λέτε κύριε Επιτρόπε ότι χρειάζεται πιο αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτή η ιστορία δεν ε, πρόκειται να σταθεί εκτός ε, και αν ε, πιο συχνά ανακοινώνουμε, μάλλον κάνουμε κάποιους μη ανακοινωμένους ελέγχους και έχουμε και κυρώσεις για μένα. το θέμα των ελέγχων πρέπει να το δούμε γιατί τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους και για τις κυρώσεις και δεν θα το επιλύσουμε αυτό το θέμα εκτό και αν βρούμε μια μαγική λύση που νομίζω ότι στην περίπτωση τη απαγόρευση των κλοβών δεν έχουμε βρει ακόμη. Εγώ θα ήθελα να έχω αποτρεπτικέ ε, κυρώσει ε, και ελέγχου έτσι ώστε να χτυπήσουμε όσου δεν σέβονται του κανόνε ε, και καταστρέφουν την κατάσταση για όλου του υπολείπου. Θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό γιατί πιστεύω ότι δεν έχουμε βρει ακόμη την μαγική λύση. Τώρα, η ερώτηση που έχω για σας σήμερα αφορά ένα νέο θέμα, το ότι ε, λαμβάνω όλο περισσότερες πληροφορίες για το ότι γίνονται απάτες κατά την παραγωγή τροφίμων. Τώρα, αν αυτό συνδέεται με την οικονομική κρίση, ότι δηλαδή υπάρχουν περισσότερες οικονομικές πιέσεις στους παραγωγούς τροφίμων, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά πολλοί εμπειρογνώμονες μου λένε ότι έχουν την εντύπωση ότι η τάση απάτης αυξάνεται κατά την παραγωγή των τροφίμων. Έχουμε το βιομηχανικό άλλα σε να καταλήγει σε πολλέ χώρε το ψωμί και στη χώρα μου και έχουμε βαρέα μέταλλα ε, και σε κάποια ε, γλυκά και μπορώ να συνεχίσω να σας δίνω τέτοια παραδείγματα που δίνουν την εντύπωση ότι τέτοιες απάτες αυξάνονται. Έτσι λοιπόν έχετε και σας την ίδια εντύπωση πόσες οι δικές σας υπηρεσίες εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές μας είναι τόσο προστατευμένοι σε μια οικονομική κρίση όταν είναι οι τιμές υψηλέ για τα εργοστάσια και τους παραγωγούς τροφίμων ή αυτές τις μέρες εργάζεστε επιπλέον ε, σκληρά για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριο Καρόνα και μετά Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του κυρίου Επιτρόπου που τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ και για τη διαθεσιμότητά του στο εξή. Τον ε, Ιανουάριο φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία ε, κατόπιν πρωτοβουλίας και αυτής της Επιτροπής ενέκρινε ένα ψήφισμα για το θέμα της κατασπατάλησης των τροφίμων. Ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρει πάρα πολλές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων και μία κατεπίγουσα, ότι το 2014 θα θεωρηθεί το, θα έχουμε μάλλον το ευρωπαϊκό έτος κατά της κατασπατάλησης ε, των τροφίμων. Ε, καθώς η απήχηση αυτού του ψηφίσματος είναι πολύ μεγάλη στις διάφορες χώρες υπάρχει και μια μεγάλη αναμονή και προσδοκία για τις αποφάσεις ή τις μη αποφάσεις που θα λάβει η Κομισιόν. Επίσης να σας ενημερώσω ότι μεταξύ άλλων σε διάφορα κοινοβούλια δραστηριοποιούνται διάφοροι βουλευτές για να αναπαράξουν σε εθνικό επίπεδο το ίδιο αίτημα. Έτσι λοιπόν, εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω πολύ μεγάλη αγωνία για να μάθω αν ε, υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από δική σας πλευρά, αν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της Κομισιόν, ε, έτσι ώστε το 2014 να μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιο ευρωπαϊκό έτος. Αυτό είναι το πρώτο ε, μήνυμα. Βέβαια, συνέχεια υπάρχουν και μία σειρά οδηγιών που θα πρέπει, μία σειρά δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν, αλλά όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε εν καιρό. Ευχαριστώ κυρία Καρόνα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ρωτήσω για το χρονοδιάγραμμα δύο συγκεκριμένων πακέτων νομοθεσίας τις οποίες περιμένουμε με ανυπομονησία αλλά έχουν καθεστήριση. Το πρώτο είναι η το πακέτο κτηνιατρικών μέτρων Μα είπαν ότι θα δούμε τις προτάσεις του χρόνου, το πρώτο εξάμεινο του χρόνου. Αυτή είναι μια μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά γιατί έχει παρουσιαστεί. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτή η νομοθεσία βασίζεται σε ένα πολύ παλιό νομοθετικό πλαίσιο και έχει άμεσο αντίκτυπο για τις μικρότερες χώρες. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε προσπάθειες να ε, ε παρουσιαστεί αυτή η νομοθεσία νωρίτερα. Ε, το δεύτερο φορά το πακέτο φυτογειονομικών ε, μέτρων υγείας ε, φυτών και ζώων, πολλαπλασιαστικό υλικό και όλα τα συναφή. Και πάλι το πακέτο αυτό καθυστερεί όσον αφορά την, τα νομοθετικά μέτρα, την νομοθεσία. Υπάρχει λοιπόν στις προτάσεις σας αυτό το θέμα. Και στα δύο αυτά θέματα λοιπόν θα ήθελα να ενεργήσετε ταχύτερα και να αντιδράσετε ταχύτερα. Περιμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Κυρία Γκαρσία, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κάποιε σύντομε ερωτήσει από τη σκοπιά τη ευζοία των ζώων. Θα ήθελα να μου πείτε αν εσεί θεωρείτε ότι ολογείται ένα τόσο αυστηρό περιορισμό, 8 ώρε μόνο για τις ε, μεταφορές στο σφαγείο, που δεν, κάτι που δεν εφαρμόζεται ε, σε κάποιες διαδρομές στη μεταφορά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτό εφαρμόζεται μόνο για τις διαδρομές προς το σφαγείο και όχι στις διαδρομές ε, τις υπόλοιπες. Και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αν το εφαρμόσουμε μόνο για τα σφανεία, θα αφήναμε εκτός τη εφαρμογής της οδηγίας το 60% των διαδρομών. δεύτερη ερώτηση. Εσείς έχετε σκεφτεί να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία στον τομέα των φυτογεωνομικών. Σα το λέω γιατί αναμένουμε από τι 14 Δεκεμβρίου πέρσι μία τεκμηρίωση, μία νομοθετική πρόταση σε σχέση με τις ίσονο σημασία ε, χρήση στο φυτογειονομικό τομέα. Και αυτό σα το λέω σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών ε, ε, φάνηκε ότι όσοι καλλιεργούν εσπεριδοειδείς στην Ευρώπη βρίσκονται σε εντελώ ανισπεράσπιστη θέση γιατί δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να του προστατεύει από τις ίσονος χρήση. χρήσης. Και τέλο, μία σύντομη ερώτηση για τη νέα νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα, novel food και για την κλωνοποίηση. Έχετε την πρόθεση να παρουσιάσετε αυτές τις δύο νομοθετικές προτάσεις ταυτόχρονα ε, ή θα έχουμε διαφοροποίηση από τη, τις κλωνοποίησεις από τα νέα τρόφιμα και θα υπάρχει δηλαδή και διαφοροποίηση κατά την εξέταση από το Κοινοβούλιο. Η κυρία Πόλσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Νταλή που ήρθε εδώ και απάντησε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σε σχέση με τον κανονισμό για, την, για τη υγειονομικά μέτρα και τα μικρά σφαγεία, ο κανονισμός θεωρώ εγώ ότι ίσως είναι παρκώς ευέλικτος ε, και το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το κόστος και ο επιμερισμός του κόστος. Όταν ε, πραγματικά ε, δέχονται δυσμενέστερη σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταχείριση τα μικρά σφαγεία σε σχέση με τα μεγάλα. Νομίζω λοιπόν ότι από πλευρά Κοινοβουλίου και Επιτροπή αλλά και Συμβουλίου αυτό πρέπει να μα επισχολήσει. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε σε λειτουργία πολλά τοπικά και περιφερειακά μικρά σφαγεία. Ε, τώρα, σε σχέση με τη στρατηγική και την πολιτική για, την, ε, για το ευζήν των ζώων, ε, ε, εξυπακούεται ότι ο έλεγχος και η συμμόρφωση είναι αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο, διότι... δεν έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη. Πάντως είμαστε πεπισμένοι ότι αν έχουμε ένα νόμο πλαίσιο όπως ακριβώς έχουμε για τα τρόφιμα δηλαδή, Πιστεύουμε ότι όλα θα ήταν πολύ απλούστερα, δηλαδή ένα απλό πλαίσιο που προσδιορίζει τις αρχές ε, για την φροντίδα των ζώων, ε, όπου ξέρουμε ποιος ευθύνεται γιατί και ποιος λογοδοτεί, ε, είναι κάτι που θα διευκόλυνε τα μάλλα και τη συμμόρφωση και τους ελέγχους. Για τους ελέγχους ε, συγκεκριμένα, σε αυτή την στρατηγική που θα ψηφίσουμε εντό ολίγου, ε, βλέπουμε ότι προτείνονται διάφορα ορόσημα. Αν έχουμε παραδείγματος χάρη μία πενταετή ή δεκαετή μεταβατική περίοδο για να αλλάξουμε οποιοδήποτε κανόνα ε, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα, δύο, τρία σημεία να ζητήσει ξεκάθαρες απαντήσεις σε σχέση με την πρόοδο που σημειώνεται σε κάθε κράτος μέλος ε, και είναι γεγονός ότι ούτως ή άλλως είμαστε δεσμευμένοι, ε, αλλά από την ημερομηνία θέση σε εφαρμογή και μετά και όχι νωρίτερα. Οπότε χρειαζόμαστε ε, λεπτομερέστερη ρύθμιση, αλλά σε προηγούμενο στάδιο, πρωτού δημιουργηθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πάουλσεν. Ο κύριος Τόρφμαν τώρα. Grazie signor Commissario. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταφοράς των ζώων, υποστηρίζω τη θέση σα γιατί είμαι πεπισμένο ότι η ευημερία των ζώων κατά τη διάρκεια των μεταφορών είναι ένα θέμα χρόνου, αλλά είναι και θέμα ποιότητα ε, της μεταφοράς. Σε όλη αυτή τη συζήτηση συχνά ξεχνάμε ότι όταν μεταφέρουμε, ότι μεταφέρουμε ένα ζώο 10-12 ώρες, το να το περιορίσουμε στις 8 ώρες σημαίνει ότι ε, ε, μπορεί να το μεταφορτώνουμε, παίρνουμε το σχάρι, να το πετάμε το ζώο. Έτσι λοιπόν τελικά δεν βελτιώνεται η ποιότητα της μεταφοράς. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε κάτι που αφορά τη χώρα μου, την Ιταλία. Ε, θέλω να αναφερθώ στο θέμα της ε, καταπολέμησης ε, της λοιπόν της γνώσης του κατά των μελισσών. Στην τελευταία έκθεση που υλοποιήσαμε για την ευημερία των μελισσών αναφερθήκαμε στο ότι χρησιμοποιούνται κάποια οργανικά οξέα. Στην Ιταλία υπήρξε ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με τη χρήση του οξέους αυτού. Ε, γιατί ποτέ δεν ε, έχει καταγραφεί ε, αυτό το οξύ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται πλέον για την καταπολέμηση θέλω, ε, αυτής της νόσου των μελισσών. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε επίγνωση αυτού του θέματος και πώς θα μπορούσε να επιληθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Ράινερς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που ήρθατε και πάλι σε εμά. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν πολύ επικοδομητικό διάλογο. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον για τα αντιβιωτικά και τη χρήση τους. Είπατε ότι θα πρέπει να είναι παρόντες οι κτηνίατροι για να δοθούν τα αντιβιωτικά στα ζώα. Πολύ ωραία το ακούγεται αυτό, αλλά πώς γίνεται τώρα να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ε, την παρουσία κτηνίατρου ιδίως ε, στα μεγάλα ζώα και όταν η παραγωγική μονάδα είναι μεγάλη ε, θα είναι τεράστιο το κόστος να μπορέσει αμέσως να αποσταλεί και να υπάρχει κτηνίατρος. Ε, τα, τα μεγάλα ζώα, τα βοηδή ας πούμε, είναι διαφορετικά από τα κοτόπουλα και τις ε, όρνησες. Ε, έχουν πόνους, δεν εμφανίζεται αμέσως το πρόβλημα, ιδίως στη μαστίτιδα. Λοιπόν, τα προβλήματα εκεί που θα προκύψουν είναι τεράστια. Και αυτό το, το οποίο έχουμε ακούσει τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι στις, ε, στα αυγά ελεύθερης βοσκής παρουσιάζονται ε, προβλήματα όχι μόνο στη χώρα μου αλλά και σε άλλες χώρες. Πώς λοιπόν θα διαχειριστούμε αυτά το, το πρόβλημα των ε, κατοφλίων ε, παροχής αντιβιωτικών έτσι ώστε παρόλο που υπάρχουν ορισμένες, ορισμένα όρια στη χρήση που δεν είναι βλαβερά για τον άνθρωπο τουλάχιστον για τα ζώα η μεταχείριση είναι διαφορετική ε, ε ως Σον, που πολλές φορές ε, επίσης πρέπει να δούμε τις συνθήκες εκτροφής των ζώων, ιδίως στα και στα κοτόπουλα, όπου τα κοτόπουλα θεωρούνται ελεύθερης βοσκής, χωρίς να έχουν όμως επαφή με το έδαφος. Ευχαριστώ κυρία Γιούσο, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τις εξηγήσεις μας. Ε, Ξέρετε τις ανησυχίες μας, γιατί σας τα έχουμε ξαναπεί, αλλά έχουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία για την ευημερία των ζώων, για τα παρασιτοκτόνα, για τους γαματαφόμητρων, για την κλωνοποίηση, για τα νέα τρόφιμα, αλλά αυτό συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα όσα εισάγουμε δεν σέβονται την νομοθεσία. Ε, δηλαδή, ε, παρόλα αυτά εμεί εισάγουμε προϊόντα που είναι πιο φτηνά ε, να παραχθούν και δεν σέβονται την ομοθεσία τη δική μας. Ε, Παραδείγματο χάρη υπάρχει έκθεση τη ΕΦΣΑ τη 4 η Απριλίου όπου αναγνωρίζεται ότι τα προϊόντα που εισάγονται από 6 έω 15 φορέ περιλαμβάνουν περισσότερα παρασιτοκτόνα από αυτά που χρησιμοποιούνται στα δικά μα προϊόντα και εδώ δεν μπορούμε εμεί ε, να καλλιεργήσουμε πάρα πολλέ καλλιέργειε, αλλά τελικά τα εισάγουμε αυτά τα τρόφιμα. Παραδείγματο χάρη, καταναλώνουμε αυγά από ορνηθε που βρίσκονται σε κάποιου κλοβού 350 εκατοστών, ενώ εμεί εδώ ζητάμε το διπλάσιο. Ε, 700 ε, εκατοστά. Εγώ σας ρωτώ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει μια εκστρατεία για να εξηγήσει στους ε, Ευρωπαίους καταναλωτές ε, ότι τα προϊόντα μας είναι πιο ακριβά γιατί είναι τα καλύτερα και γιατί δεν ζητάμε τα προϊόντα που δεν σέβονται τους μα κανόνε να μην μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να βρει κάποιο ένα προϊόν που δεν σέβεται την νομοθεσία και να κλείσουμε τα σύνορα στη χώρα αυτή και μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε και του δικού μα γεωργού. Ε, έχω κάνει και μια γραπτή ερώτηση για αυτά τα δύο θέματα και μου απαντήσατε κάτι άλλο. Και τώρα δράτω την ευκαιρία να σα πω να πείτε στου υπαλλήλου σα να απαντούν σε μια ερώτηση, να απαντούν σε αυτό που ρωτάμε όχι σε, να ξεφευγούν από το θέμα. Σας ευχαριστώ, δεν θέλω να χάσουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Νικολέσκου. Pan poseł Nikolescu takim razie επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικό που αναφέρθηκε πριν την αθεώρηση της οδηγίας ε, για τα προϊόντα καπνού. Με ικανοποίηση σα άκουσα να λέτε σήμερα το απόγευμα ότι η αναθεώρηση αυτή τη οδηγία ε, δεν θα αφήσει δραστικά του γεωργού. Όμως κατά την άποψή μου η αναθεώρηση αυτής της οδηγία ε, θα σημαίνει ένα ισχυρό πλήγμα για την καλλιέργεια και την παραγωγή καπνού ενός τομέα που δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας ε, σε ζώνες ε, που βρίσκονται ε, στο στόχο σύγκλησης όπου το ποσό της ανεργίας ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Το τομέας αυτός είναι μια πολύ σημαντική πηγή απασχόλησης όπως συμβαίνει στην Εστραμαδούρα παραδείγματος χάρη όπου δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ παραγωγές. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει διόντως υπόψη τις δραστικές αλλαγές που θα μπορούν να επιφέρει αυτή η αναθεώρηση για όλους όσους συμμετέχουν στην παραγωγή, στην εμπορία και για τον καταναλωτή στην Ευρώπη. Κύριε Επίτροπε, δεν πιστεύετε ότι θα ήταν απαραίτητο να εισαχθεί ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σταθερό ε, και να βασιστούμε σε ε, παρκή αξιόλογα επιστημονικά στοιχεία που θα μπορούσαν ε, να έλθουν σε αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Πίτροπος πρέπει να φύγει στις 4.30. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους επόμενους να είναι τηλεγραφικοί. Θα είμαι αρκετά σύντομος και θα μιλήσω για το γενικότερο πλαίσιο. Όλες οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση του τέστην προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, της διευκόλυνσης. Αυτό που όμως που με ξαφνιάζει εμένα είναι ότι ταυτόχρονα επανεθνικοποιείται ο διάλογος ε, και τίθε το ενδεχόμενο να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε τους κινδύνους ε, που εγκυμονεί αυτό για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι ευρωπαϊκός ο διάλογος για να έχουμε έχουμε πραγματική ουσιαστική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι επικίνδυνο λοιπόν να θέλουμε να επιστρέψουμε στο εθνικό πλαίσιο. Βλέπουμε με τα παρασιτοκτόνα τι γίνεται παραδείγματο χάρη. Έχουμε την νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην αμπελουργία όμω ε, και στου ε, λάχανόκηπου στα απορροκυπευτικά, μεγάλη χρήση παρασιτοκτόνων. Οπότε προσοχή κρού τον κόδωνα του κινδύνου, α μην ξαναγίνουν εθνικέ συζήτησει για αυτά τα ζητήματα. Πρώτον. Δεύτερον, την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρετε ότι προβλέπεται ψηφοφορία για το θέμα του αν θα δεχτούμε ε, τους λογαριασμούς ε, της αρχής ε, τροφίμων, ασφάλεια των τροφίμων, της ΕΦΣΑ. Γιατί, διότι υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων, συζητήθηκε το θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και προτείνει η Επιτροπή Κόντ, λοιπόν, να καταψηφίσουμε τους λογαριασμού λογαριασμού του οργανισμού αυτού. Αν έχει φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο, πάει να πει ότι σε διάφορα βήματα δεν έχουμε διαφάνεια και άρα δεν πρέπει ανα αναδιαρθρώσουμε αυτόν τον οργανισμό, τόσο ώστε να είναι διαφανής. Δεν είναι ότι υπήρξε οποιαδήποτε υπεξαίρεση, κατάχρηση ε, και το καθεξή αλλά δεν εργάζεται ο ε, οργανισμός πλέον όπως θα έπρεπε και δεν καλύπτει πλέον ούτε τι ανάγκε για διαφάνεια που ζητάει το Κοινοβούλιο δηλαδή, ούτε ε, καλύπτει τις ε, προσδικίες των κρατών μελών. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα επιστημονικά μας στοιχεία για να κάνουμε μια εις συζήτηση. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να δοθεί η απαλλαγή από το Κοινοβούλιο στον ΕΦΣΑ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νταντάν τώρα... Ε, όχι, Ευχαριστώ. δύο ίσονο σημασία ερωτήσεις, γιατί τα, με πρόλαβαν οι συνάδελφοι για τις καλλιέργειες προβλέπετε να κάνετε πιο αυστηρή την νομοθεσία για τα ε, χωροκατακτητικά είδη ε, ε, όταν η εμπορία τους όμως, όταν εμπορευματοποιούνται ως καλοπιστικά ε, τίθεται μεγάλο πρόβλημα ε, για την φύση. Απειλούνται άλλα είδη. Τώρα, σε σχέση με το περιθώριο του πακέτου για τα υγειονομικά μέτρα, υπήρχαν διατάξεις για τους μικρούς ε, παραγωγούς που εφαρμόζουν τη μέθοδο της άμεσης πώλησης. Υποθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούμε να έχουμε ένα συλλογικό έγγραφο με τις διατάξεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ακούσαμε αυτή την πρόταση, αλλά οι γεωργοί που ασχολούνται με τις άμεσες πωλήσει, παρόλα αυτά θεωρούν ότι ε, είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες. Ε, θα τους καταστήσετε ελαστικότερους. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ποζεχόφσκι και η κυρία Γκέρι. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο με ανησυχεί λίγο η θέση σας στο θέμα της μεταφοράς των ζώων όπου απορρίπτεται ξεκάθαρα το όριο των 8 ώρων ή εν πάση περιπτώσει απορρίπτεται κάθε όριο χρονικό όριο μεταφοράς. Πράγματι, είναι δαπανηρή μεταφορά των ζώων και το υψηλό κόστος αυτό αντανακλάται συνεχεία στο, στις λιανικές τιμές και επιβαρύνει τους καταναλωτές ε, αλλά το κόστος ε, κάπου θα πρέπει να πέσει. Ε, είναι όμως γεγονός ότι πολλές φορές οι μεταφορές είναι πολύ περισσότερο από 8 ώρες μέχρι και 24 ώρες και πάρα πολύ ακριβές. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η μεγάλη πίεση και από πλευράς ε, καταναλωτών επιβληθεί ένα τέτοιο όριο αλλά και από τις διάφορες περιφέρειες ε, υπάρχει πίεση. Εάν μπει ένα τέτοιο όριο θα πρέπει να υπάρχουν και περισσότερα σφαγεία, περισσότερες εγκαταστάσεις σφαγής. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις ε, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι εύλογο να βρούμε ένα όριο, ένα συμβατό όριο μεταφοράς, ε, διότι αντίθετα ε, από τις προθέσεις της Κομισιόν, ο κανονισμός λέει ότι θα καταλήξει τελικά σε, μία, σε ένα όριο, σε μία μείωση των, του χρόνου μεταφοράς. Ενώ αυτή τη στιγμή το μήνυμα έρχεται, που έρχεται είναι εντελώς αντίθετο. Αντί λοιπόν να απορρίψετε αυτή την πρόταση θα πρέπει να την ξαναμελετήσετε. Ευχαριστώ κυρία Γκέρλινγκ. Θα είμαι όσο πιο σύντομη μπορώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντάλι που ήρθε σε εμάς δεν θα σας ζητήσω συγγνώμη που θα επαναλάβω κάτι που είπα και προηγουμένως και αφορά τις επιστημονικές ενδείξεις για τις ε, συγκεκριμένες συνθήκες μεταφοράς αλόγων, υπο, ύπων, και υποειδών. Δεν έχει γίνει καμία συγκεκριμένη συζήτηση για τις ειδικέ συνθήκες μεταφοράς ύπων και υποειδών Είχαμε ε, μέσα στα πλαίσια της ΕΦΣΑ συζητήσει το θέμα αυτό και είχαν συμφωνήσει ότι έχουν ιδιαιτερότητες τα άλογα και τα υποειδή και γι' αυτό θα σας παρακαλούσα ειδικά για την κατηγορία αυτή των ζώων να σκεφτείτε την, το περιορισμό των 8 ωρών. Ε, εντάξει, δεν λέω ότι οριζόντια θα πρέπει να επιβάλλουμε τις 8 ώρες, αλλά υπάρχει πληθώρα επιστημονικών ενδείξεων που λένε ότι αυτό το όριο πρέπει να επιβληθεί στους ύπους και στα υποειδή. Ιδιαίτερα όταν μεταφέρονται πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός των συνόρων στα Ανατολικά. Αυτό πραγματικά πρέπει να σταματήσει. Επίσης, υπάρχει διαφορετική ερμηνεία ε, στα θεσμικά όργανα. Εγώ από ό,τι κατάλαβα η Δανική Προεδρία απέριψε κάθε περαιτέρω διαβούλευση στο πακέτο των γενετικά τροποποιημένων. Η διαδικασία συνδιαλλαγής όμως δεν συνάδει με ε, αυτό το οποίο έχω ακούσει και γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω αν το πακέτο των τροποποιημένων θα συζητηθεί στο Συμβούλιο ή όχι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει τον τελευταίο γύρο των ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις απάτες στα τρόφιμα. Δεν γνωρίζουμε να υπάρχει δραματική αύξηση στις απάτες στα τρόφιμα. Σας δώσω ένα παράδειγμα αυτό το περιστατικό που αναφέρθηκε πρόσφατα για τα βιομηχανικά άλατα σε παραγωγή κάποιων τροφιμών από την Πολωνία που εξαγάγονταν στη Τσεχία. Από ό,τι φαίνεται λάμβανε χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς τώρα το μάθημα δεν ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω ότι πρέπει συνεχώς να επαγρυπνούμε για να ελέγχουμε και να καταπολεμούμε την απάτη. Δυστυχώς, η απάτη είναι κάτι που θα συνεχίσει να μας πλήττει. Όχι μόνο στην παραγωγή των τροφίμων, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Και δεν μπορούμε παρά να αποδηγήσουμε κάθε πέτρα για να καταπολεμήσουμε την πρακτική αυτή. Για τα πόβλητα τροφίμων. Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον συνάδελφο, τον Επίτροπο Ποτότσνικ, ε, για το θέμα των υποβλήτων ε, της πατάλης των τροφίμων και αναμένουμε να υπάρξει και μία ανακοίνωση πολύ σύντομα για το θέμα αυτό. Η σπατάλη των τροφίμων είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κάθε πολίτη ε, στην Ευρώπη παραγεί 180 κιλά ε, τέτοιων αποβλήτων ετησίω ε, και πρόκειται πραγματικά για σπατάλη. Έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και έχει και μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία. Και είναι ένα ζήτημα με πολλές πτυχές. Εγώ συμμετείχα σε μια διάσκεψη με τον κύριο Ποτότρινγκ πέρσι για το θέμα αυτό όταν ε, συμμετείχαν και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και πραγματικά ασκούμε πίεση για να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση και μια καλύτερη εκπαίδευση των πολιτών μας για το θέμα αυτό. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφοροποίηση στην ετικοθεσία των ε, τροφίμων ε, σε σχέση με την ημερομηνία λήξη. Καλύτερα να καταναλωθεί μέχρι τότε ή πρέπει να καταναλωθεί μέχρι την τάδη ημερομηνία. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα, η ημερομηνία λήξη είναι ένα θέμα υγεία. λέμε ότι μην το χρησιμοποιήσετε, μην το καταναλώσετε μετά από μια ημερομηνία, αλλά το best use before ότι καλό θα ήταν να καταναλωθεί μέχρι τότε, απλώ αναφέρει ότι μετά από κάποια ημερομηνία αλλοιώνονται κάποιε από τι ποιότητε. Ε, κάποια από τα συστατικά. Μπορεί να καταναλωθεί όμω ακόμη το τρόφιμο και ήδη με κάτι τέτοιο θα εξοικονομούσαμε πολλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, ε, κατά το πρώτο εξάμεινο του 2013 σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε νομοθετικές προτάσεις. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που πιστεύουμε ότι είναι πρακτικό να θέσουμε ως στόχο επίσης γιατί θέλουμε να το συνδυάσουμε και με τις ε, προτάσεις μας για την ε, αντιμικροβιακή αντίσταση. Επίσης, μας ενδιαφέρει να δούμε αν ε, μπορούμε να δώσουμε κάποια παρότριση και εργαζόμαστε με τον κλάδο σε αυτό το τομέα, μπορούμε να δώσουμε κάποια παρότριση στο να αναπτυχθούν ορισμένα κτηνιατρικά εμβόλια που θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιηθούν ε, στα ζώα και όχι στους ανθρώπους. Και εργαζόμαστε και από αυτού λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταφορές και πάλι, τη μεταφορά των ζώων, το θέμα είναι να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες επιστημονικές ενδείξεις, περισσότερα επιστημονικά στοιχεία Τώρα το μελετώ εις βάθος ε, το θέμα και στο παρελθόν, αλλά και τώρα εξακολουθώ να αμφισβητώ την ανάγκη για τη μεταφορά, λέγοντας ότι κάποιες φορές πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της ετικέτας προέλευσης ε, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, γιατί χρειάζεται πολύ, μεγάλη μεταφορά. Τώρα όμως αφενός, αν σκεφτεί τι συμβαίνει και ε, πώς έχει να διερθρωθεί ο κλάδος ε, στην Ευρώπη, έχει γίνει μεγάλη αναδιάρθρωση, τα σφαγεία γίνονται ένα και μεγαλύτερα. Ακούσαμε εδώ ε, ότι κλείνουν ε, τα μικρά σφαγεία. Εγώ δεν συμφωνώ απαραίτητα με κάτι τέτοιο, αλλά αυτό συνέβη τα τελευταία έτη. Και να προσπαθήσουμε τώρα να αντιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία δεν είναι κάτι που μπορεί να ε, το δούμε απλά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί Δηλαδή, ναι μεν ε, υπάρχει ιδανική κατάσταση, αλλά πρέπει να δούμε και τι είναι δυνατόν εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σόφρον να έχουμε νέους ειδικού κανόνες ε, για ε, τη μεταφορά των ζώων. Επιτρέψτε μας να επικεντρωθούμε στην επιβολή της νομοθεσίας και να επιβάλλουμε την νομοθεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μας επιτρέπει η σύγχρονη τεχνολογία. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. για τη συμβουλή της κυρίας Πόλτσε να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο για την ευημερία των ζώων. Αυτό ακριβώ κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ε, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος και για να εισαγάγουμε κάποια ευελιξία στο πώς ε, εξετάζουμε την ευζοία των ζώων και να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα παρά στις συγκεκριμένε διαδικασίες. Αυτό θέλουμε ουσιαστικά να πράξουμε. Σε ό,τι αφορά τι μεταβατικέ περιόδου, και πάλι συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, ε, νομίζω ότι δημοσίω είναι γνωστό ότι πρέπει να μάθουμε από τις εμπειρίε που πρόσφατα είχαμε και είχα και εγώ σε σχέση με τις οτόκες όρνηθες. <coughs> Η μεταβατικές ε, διαδικασίες ε, είναι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα όμως, αλλά αν έχουμε αυτές τις διαδικασίες, σας διασφαλίσουμε ταυτόχρονα ότι καλύπτονται και από ε, την εφαρμογή. Δηλαδή, κάθε, κάθε, σε κάθε κράτος μέλος να μπορεί η Κομισιόν να ελέγχει ότι υπάρχουν προγράμματα εφαρμογής τα οποία γίνονται σεβαστά. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τελικά θα έχουμε εφαρμογή σε όλες τις χώρες. Και ίσως ε, τότε, ε, αν η Κομισιόν δεν έχει αναλάβει δράση, τότε να την κατηγορήσετε. Η Κομισιόν δεν μπορεί να δράσει πριν τη λήξη της μεταβατικής περίοδου είναι εντελώ δεμένα τα χέρια μας. Τώρα, για τις μέλισσε. Και για τα, αντιμικρο... για τα αντιμικροβιακά, με συγχωρείτε. Όταν ενημερωθήκαμε για τις εκθέσεις αυτές, αναλάβαμε όμως τη δράση, στείλαμε τις εκθέσεις στην ΕΦΣΑ για να κάνει μια συγκεκριμένη ανάλυση, στοχευμένη ανάλυση των εκθέσεων αυτών για να μελετήσει τη δοσολογία. Αν ε, η δοσολογία που χρησιμοποιούνταν στο εργαστήριο όπου έγιναν ε, οι εκθέσεις είναι οι ίδιες δόσεις που χρησιμοποιούνται και στους αγρούς και αναμένουμε την έκθεση της ΕΦΣΑ πολύ σύντομα. για τη διοξίνη, για τα αυγά. Τα κράτη-μέλη είναι πολύ βέστητα για το θέμα αυτό. Προγράμματα, αυστηρά προγράμματα ελέγχου εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη-μέλη. Το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Είχαμε την περίπτωση της Γερμανίας ε, με τη διοξίνη πέρσι και μπορώ να πω ότι όταν ενχνεύτηκε αυτό υπήρξε ταχεία ανάληψη δράσης από τη Γερμανία και πράγματι πολύ σύντομα τέθηκε η κατάσταση από έλεγχο. Σε σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων, από άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η κυρία Γιούσο το έθιξε. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την ευζοία των ζώων ε, ως ε, μέθοδο υπερασπισή μας εμπορικής άμυνας. Έτσι λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση στο όσα είπε η κυρία Ιούσο και συμφωνώ πολύ μαζί τη ότι οι δικές μας πολιτικές για την ευζοία των ζώων δεν είναι απλώς ένα θέμα ευημερία των ζώων κάτι στο οποίο πιστεύουμε είναι θέμα και ποιότητα των τροφίμων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ζητούν οι πολίτες για τα προϊόντα καπνού. Και πάλι, είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλές θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτό και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι το λαμβάνουμε απολύτω υπόψη αυτό στη μελέτη αντικτύπου που προετοιμάσαμε. Παρ' όλα αυτά, ο καπνός ε, προκαλεί και θανάτους. 650.000 άνθρωποι ετησίως πεθαίνουν λόγω του καπνίσματος και είναι μεγάλη απώλεια αυτή και οικονομική. Πέρα από το τι υποφέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι και μεγάλη οικονομική απώλεια. Και υπάρχει και μεγάλη πίεση στην ε, βιωσιμότητα των ε, υγειονομικών συστημάτων. Τώρα, σε σχέση με τους ε, γενετικά τροπομένους οργανισμούς εδώ, και πάλι, η Επιτροπή ανέλαβε δράση κατόπιν αιτήματος 12 κρατών μελών θεωρήσαμε ότι αυτή η πρόταση ήταν βιώσιμη. Είναι βιώσιμη γιατί η γεωγραφική κατάσταση, η κατάσταση επιμελητία σε διάφορα κράτη-μέλη ζητούν να ληφθούν συγκεκριμένε αποφάσει από κάθε κράτο μέλο ό,τι αφορά την καλλιέργεια των γαμματα δεν πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί πράγματι προβλήματα για το αν καλλιεργούνται ε, περισσότερο γαματαφό Στην Ευρώπη όχι. Δεν ε, είναι θέμα αν θα επανέλθουν οι γαματαφό μικρών ή αν έφυγαν. Το θέμα ε, μας απασχολεί, υπάρχει και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και στο μέλλον, καθώς η Ευρώπη θα δέχεται όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση και η ανάπτυξη στην παραγωγή γαμματά όμικρον ε, σε άλλε χώρε ε, θα αυξάνεται. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και θέλω να απευθύνω έκκληση σε όλου να το αντιμετωπίσουμε αυτό αντικειμενικά και λογικά. Λαμβάνοντα υπόψη όλα τα θέματα ασφάλειας και όλα τα περιβαλλοντικά θέματα. Όπως γνωρίζετε, όταν ε, άρχισα να ασχολούμαι με τα θέματα αυτά, είχα δηλώσει ότι είμαι υπέρ της καινοτομία, αλλά υπέρ της υπεύθυνη καινοτομία. Και η υπεύθυνη καινοτομία διασφαλίζει την ασφάλεια και το φέλη της κοινωνίας. Και αυτό προωθούμε αυτή τη στιγμή γιατί η διαφάνεια της ΕΦΣΑ. Να πω ότι έχουμε κάνει πολλά είδη στην ΕΦΣΑ για να διασφαλίσουμε την διαφάνεια από την αρχή ε, της σταδιοδρομίας μου εδώ ακούω τα θέματα αυτά και εξακολουθώ να σκοπίεσαι για να συνεχίσουμε να προωθούμε τα θέματα της διαφάνειας στην ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ ήδη έχει λάβει πολλά μέτρα για να ελέγξει όλους όσους ενέχονται στις επιστημονικές αξιολογήσεις. Έχουμε προβλήματα ενίοτε. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Αλλά και πάλι εδώ σας διαβεβαιώ ότι αναλαμβάνουμε δράση και επιμένουμε ως Επιτροπή στην άμεση ανάληψη δράσης. Βέβαια, έχουμε κατά νου ότι είναι αυτόνομο όργανο η ΕΦΣΑ. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να πάω και να διατάζω την ΕΦΣΑ για το ποιος πρέπει να είναι στο Συμβούλιο και ποιος δεν πρέπει να είναι. Αλλά καθιστούμε απόλυτα σαφές ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο το θέμα της ε, διαφάνειας αυτής καθ' αυτής, αλλά και την αντίληψη της διαφάνειας, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για γεγονότα, μιλάμε και για την εντύπωση που πρέπει να έχουν οι πολίτες μας ότι όταν κάτι έχει εγκριθεί από την Εύσα, έχει εγκριθεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Συμφωνώ με αυτό. Και όπως ξέρετε, πάντοτε είναι πρόσδεκτα τα σχόλιά σα για οποιαδήποτε δράση μπορούμε να λάβουμε προ αυτήν την κατεύθυνση, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε. Ε, ε- Μετά, ξένα ήδη. Of pesticides Um, πεταλοδαπά και χώρο επεκτατικά. Συνεργαζόμαστε με τον τομέα και τους παραγωγούς και ελπίζω ότι η έκθεσή μας για αυτά τα ε, προϊόντα θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα ε, παράλληλα και με τις προτάσεις για τα γενετικά τροποποιημένα. Το Κοινοβούλιο για τα γενετικά τροποποιημένα έχει ξεκαθαρίσει τις απόψεις του εντάξει και έχει ψηφίσει κιόλας για αυτές. Ε, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα εκδώσει απόφαση και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Το περασμένο Μάρτιο δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, δεν ξέρουμε εάν θα επανέλθουν τα γενετικά τοποποιημένα τον Ιούνιο ή όχι. Εάν επανέλθουν τον Ιούνιο θα λάβει θέση το Συμβούλιο και εν συνεχεία πρέπει να συζητηθούν αυτές οι δύο θέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου Συμβουλίου για να βρεθεί μία λύση ε, μεταξύ των δύο αυτών θέσεων. <clears throat> Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ε, έχουμε δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, για περισσότερες ερωτήσεις, αλλά ελπίζω ο κύριος Επίτροπος να επανέλθει σύντομα για μια νέα ανταλλαγή απόψεων, στην οποία προσβλέπουμε. Τον ευχαριστούμε ξανά για την παρουσία του εδώ και ένα λεπτό διάλειμμα, παρακαλώ, για να ξαναρχίσουμε. Σε ένα λεπτό. <clears throat> Proszę Państwa, przechodzimy do Θα προχωρήσουμε στις ψηφοφορίε λοιπόν. Έχουμε εδώ ε, τις ε, καταλόγους, τις λίστες. Uh,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 Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίαση για να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Η πρώτη είναι το σχέδιο έξεσης του Λούις Κάπουλα Σάντος για την τροποποίηση του κανονισμού 73 κάθετος 2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013. Διακόπτει ο πρόεδρος. Czy możemy zaczynać? Παρακαλώ, μπορούμε να ξαναρχίσουμε. Bardzo dziękuję. Λοιπόν, ξαναρχίζει η συνεδρίασή μας και Συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Επαναλαμβάνω, η πρώτη είναι ε, η ψήφιση του, της γνωμοδότησης του Λουίς Μανουέλ Κάπουλα Σάντος για την τροποποίηση του κανονισμού 73 2009 όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων ε, στους γεωργούς για το έτος 2013. Έχουμε 14 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και υπάρχουν στην, αναφέρονται στον κατάλογο ψηφοφοριών. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού έχει υποβάλει γνωμοδότησή της και προτείνει την υιοθέτηση της πρότασης της Κομισιόν, της Επιτροπής. Ε, ο εισηγητής... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ένα λεπτό μόνο. Πρόκειται για την πρώτη ψηφοφορία που θα κάνουμε σε σχέση με το πακέτο μεταρρύθμιση τη κοινή ε, αγροτικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα κανονισμό πάρα πολύ τεχνικό, αλλά που είναι θεμελιώδη, ε, γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε τη μεταβατική περίοδο. Πιστεύω ότι στις ε, προτάσεις που εγώ ίδιος παρουσίασα είτε στις τροπολογίες περιλαμβάνονται οι κύριες ανησυχίες που θα μπορούσαν ε, να τεθούν από τα διάφορα κράτη-μέλη. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι και η δική μου έκθεση αλλά και οι τροπολογίες ε, για τις οποίες ευχαριστώ θα συνεισφέρουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια μεταβατική περίοδο στο σημερινό μοντέλο και στη νέα αγροτική πολιτική. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τη Γραμματεία και την ε, Επιτροπή για κάθε υποστήριξη για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης που όπως σας είπα είναι ιδιαίτερα τεχνική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Με... Έχετε έτοιμε τις κάρτες σας παρακαλώ. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Πέρας της ψηφοφορίας. Βλέπετε στον πίνακα τα αποτελέσματα, δεν θα πω λοιπόν τι γίνεται, απερίφθη λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 11. Τροπολογία 11. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Προχωρούμε στα εκτιμώντας άρθρο 2, ε, τροπολογία 1. Όχι. Ε, α, έχουμε, έχουμε το, ε, προφορική τροπολογία της κυρίας Μαγκίνες, επί του άρθρου 1. Ε, η κυρία Μαγκίνες, αφορά τα άρθρα 68 και 69, το κείμενο δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως εδώ στο έγγραφο που έχετε στα χέρια σας, γι' αυτό θα το διαβάσω. Αφορά την παράγραφο 8 1η Αυγούστου 2012 ή ένα μήνα μετά τη δημοσίευση, τα κράτη-μέλη θα λάβουν την απόφαση που αναφέρεται στο άθρο παράγραφο παράγραφο 1 και μπορούν να την αναθεωρήσουν και να αποφασίσουν από το 2013 κλπ. Το δεύτερο είναι άρθρο 69 παράγραφο 1 και τροποποιείται ω εξή. Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν από 1η Αυγούστου 2009, 1η Αυγούστου 2010, 1η Αυγούστου 2011 ή 1η Αυγούστου 2012 ή ένα μήνα μετά την ε, ημερομηνία δημοσίευσης τη χρήση από, τη χρησιμοποίηση από το έτος που ακολουθεί την απόφαση του 10% κλπ. κλπ. Προστίθεται λοιπόν το ένα μήνα μετά τη δημοσίευση. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή ε, συμφωνεί με αυτή την προφορική τροποποίηση. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, λέει ο εισηγητή. Ευχαριστώ. Οπότε προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, το άρθρο 1, ε, πέραση της ψηφοφορίας. Δεκτή δεκτή η προφορική τροπολογία. Προχωρούμε τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, πέρας της Δεκτή. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Δεκτή. τροπολογία 14 βλέπω ότι Α, ναι, άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε τη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Δεκτή, δεκτή. Προχωρούμε στα στις νομοθετικές προτάσεις με τις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτά, δεκτή. Προχωρούμε τώρα στην ψήφιση του σχεδίου νομοθετικής γνωμοδότησης. Άρχεται, πέρας. Δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε την απόφαση να αρχίσουμε διαβουλεύσει με το Συμβούλιο μέσα στο πλαίσιο μιας συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Δεκτή. Δεκτή. Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία της έκθεσης του James Nicholson Θέλει ο συγητής να προσθέσει τίποτα πριν αρχίσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σήμερα θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση για την προαιρετική επισήμανση του βοήου κρέατος που είχε αναβληθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση διότι η Κομισιόν είχε ελαφρώς τροποποίησει την πρόταση. Οι τροποποίησεις αφορούν την ευθυγράμμιση α, και τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Η τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν είναι πιο ικανοποιητική για το Κοινοβούλιο. Έχω λοιπόν υποβάλει δύο ακόμα τροπολογίες στο θέμα των κυρώσεων μέσα στο πλαίσιο αυτής της τροποποιημένης πρότασης. Εγώ πιστεύω ότι οι κυρώσεις πρέπει να υπόκεινται στις ε, πράξεις κάτω εξουσιοδότηση, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να έχει κάποιο έλεγχο επί του θέματος αυτού στο μέλλον. Ένα λεπτό, παρακαλώ να πάρει τη θέση του ο Πρόεδρος μας. Σα ζητώ συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 23. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφορία για την 24. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφορία για την 25. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Για την 26. Άρχεται η ψηφορία. Ψήφισατε όλοι ωραία. Εγκρίνεται θα έλεγα. Άρχεται η ψηφορία. Για τις 27 και 28 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. 27 και 28 μαζί. Πέρας. Απορρίπτονται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 60. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τις 29 και 30 από κοινού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφορία για την 5. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφορία για την 31. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 32 και την 6 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Να περάσουμε στη ψηφοφορία των 34 και 35 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε την 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Να πάμε στην 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 40, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την υπαριθμόν Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί τις 36 και 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τις 39 και 41 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνονται. 43. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 44. Λέων κλπ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πενήντα. Άρχεται η ψηφορία για την 50. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφορία. αέρας Απορρίπτεται. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 62. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και η 62. Τέλος 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και ας περάσουμε στα κτιμώντας. 1. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και εκτιμώντας 11 και 12 μαζί. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 2-13 μαζί. Άρχεται η ψηφορία. 2 και 13. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται. Πάμε στην 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 3. Άρχεται η ψηφοφορία για την 3. Για το εκτιμώντας 3. Εγκρίνεται θα έλεγα. Ας περάσουμε στο 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται θα έλεγα. 59. Όχι. Άρχεται η ψηφοφορία για το εκτιμώντας 59. Και αυτό εγκρίνεται. Όχι. Είναι. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το υπερθμό 4. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 16. Συγγνώμη. Θα ψηφίσουμε το 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και 21 και 22 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και τώρα τελική ψηφοφορία για την νομοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Στον κύριο Καπλοσάντος. Όχι. Ο Σμπαλιάτο. Ακεί οι κομπλιμέντι. Στο Σέρτζο Γουτιέρε. Όχι. Oh, anyway, thank you. Τέλο πάντων, σα ευχαριστώ. Φιλάκια. Ναι, Allora, adesso colleghi, abbiamo una, una discussione. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια συζήτηση και κλεισμένων των θυρών. για τι πλέον μειονεκτικές περιοχέ. Η Κομισιόν πρέπει να μα παρουσιάσει κάποια δεδομένα. Έτσι λοιπόν, σα παρακαλώ, όσοι δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Abbiamo votato Nicholson? Sì, Λοιπόν, όσοι δεν είναι μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Έχουμε μια συνάντηση για κλεισμένο των θυρών με τα μέλη της Επιτροπής για τα μελλοντικά κριτήρια για τον καθαρισμό των πλέον μενοκτικών περιοχών. Και κλεισμένο των θυρών λοιπόν η συνεδρίαση αυτή. Μόνο οι βουλευτές μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα